πρέπει απλά με ορθές πρακτικές και με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με αυτά να δουλεύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση τώρα και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Το επόμενο θέμα είναι η προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν που αφορούν την νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις κρίση και μιμιέ. κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Το νόημα, η αφορμή για την ερώτηση αυτή ήταν οι δραστικές αλλαγές που έχουν γίνει στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μεγάλη οικονομική ύφεση την οποία περνάμε αυτή την περίοδο η αναθεώρηση της ε, πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει συγκεκριμενοποιήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση το παράνομο εμπόριο που αντιμετωπίζουν πολλές οικονομίες ε, και πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. πράγματι όλα αυτά είναι πολύ επικοδομητικά και η ερώτησή μας τώρα είναι πόσο έχουν προχωρήσει πόσα κράτη μέλη έχουν νομοθετήσει αυτές τις προτάσεις και πού βρισκόμαστε. αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια δραματική κατάσταση δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες οι οποίες παρουσιάζουν τη μεγάλη οικονομική ύφεση και αυτές είναι η ελλάδα η πορτογαλία και η ιρλανδία. παρουσιάζεται πλέον μια ταχύτατη αδυναμία εξόφλησης των δανείων που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες ο οικονομικός τους προγραμματισμός ήταν διαφορετικός η αγοραστική δύναμη των πελατών τους έχει μειωθεί με τη μείωση των μισθών κατά 50%. πρέπει λοιπόν κύριε επίτροπε εισηγούμε να γίνει μια κεντρική ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. θα πρέπει να υπάρξει μια χρονική επέκταση της αποπληρωμής των δανείων τους και επίσης εισηγούμε τη μείωση των επιτοκίων με βάση το euribor. κύριε επίτροπε η κατάσταση στις μικρομεσαίες Ευχαριστώ πολύ κυρία Τζαβέλα. Ο κύριος τώρα δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο πρόεδρος Μπαρόζο την ανέδειξε ιδιαίτερα. 99% των επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 250 εργαζομένους. Η ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά για την απασχόληση και την εκπαίδευση. Με το Small Business Act η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε μια πρωτοβουλία ώστε η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις ΜΜΕ να βελτιωθεί. Σε αυτά τα πλαίσια επίσης προβλέφθηκε και αυτό το τεστ ε, εκτίμησης επιπτώσεων για τις ΜΜΕ. Τώρα μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι η εφαρμογή αυτού του τεστ στα επιμέρους κράτη-μέλη διαφοροποιείται και πολλές φορές δεν είναι καλά τα αποτελέσματα. Μόνο πέντε κράτη-μέλη κάνουν αυτό το τεστ ΜΜΕ ε, άλλα ε, πολύ αραιά και με διαφοκειμενόμενη ποιότητα και τα υπόλοιπα δεν το κάνουν καθόλου το τεστ αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, κάναμε αυτή την επερώτηση και ζητούμε μια πρωτοβουλία από την Κομισιόν ώστε η, ε, να γίνεται αυτό το τεστ, ε, αυτή η εκτίμηση επιπτώσεων θέλουμε, η γραφειοκρατία και τα κόστη να προσδιοριστούν ποσοτικά. Θα πρέπει να διαφυλαχτούν και να προστατευτούν οι ΜΜΕ από μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που τις φορτώνει όλο περισσότερο με γραφειοκρατία και διοικητικά έξοδα. Θέλουμε η ε, εφαρμογή να γίνει ευέλικτη, να έχουν περιθώριο ελιγμών και τα κράτη-μέλη. Ο στόχος όμως πρέπει να είναι τα συμφέροντα των ΜΜΕ να λαμβάνονται υπόψη και μάλιστα με ολοκληρωμένη προσέγγιση νομοθετική. Και θέλουμε η Κομισιόν να προβάλλει να, ε, ε, υποδειγματικά τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας. Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσουμε η νομοθεσία να μπορούν να εφαρμόζονται, να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Ευχαριστώ και ο κύριε Τόιρα. Ο κύριος Μπαρνιέ για την Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, η πρώτη μου λόγη θα είναι ε, να ζητήσετε, να σας ζητήσω να συγχωρήσετε τον συνάδελφο Ταγιάννη, ο οποίο, όπω ξέρετε θα ήθελε πάρα πολύ να έρθει εδώ, διότι προσέχει πάρα πολύ αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα, αλλά έχει να προετοιμάσει την ομάδα των 20, τον G20, τον Πιθανό. Οπότε και εγώ, ω Επίτροπο Ιστορική Αγορά, ε, μπορώ αντί εκείνου να σα εξηγήσω τι θέλω να σα πει, να σα ακούσω, γιατί επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Τζαβέλα, την κυρία Τζαβέλα, την, ε, τον κύριο Τρόιρερ, γιατί με όλη αυτή την πρωτοβουλία μας ε, ζήτησαν να ξεκαθαρίσουν τι θα γίνει με το νομοθέτημα για τις ΜΜΕ ε, και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα 20 εκατομμύρια των επιχειρήσεων που είναι 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίοι κατά 90% δημιουργούν ναι, την απασχόληση 90% γιατί μιλούμε πάντοτε για μη μη ε μιλούμε για για ε, το 90% του, του, του οικονομικού ιστού της Ευρώπης. Μιλούμε για το κλειδί για την ανάπτυξη που θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε, δυναμισμό στην οικονομία, ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά τα οποία θέλουμε, για αλλά όμως έχουν τώρα όλες αυτές οι επιχείρησεις ιδιαίτερες δυσκολίες ε, τη σήμερα ημέρα, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα οι ΜΜΕ πάρα πολύ σημαντικούς φραγμούς στην πρόοδό τους, οι οποίοι συνεχίζονται όσον αφορά κινητικότητα για τις εξαγωγές, για τις ενταλλαγές πέραν των ε, μεγάλων αγορών και όλα αυτά θα ήθελε ο κύριος Σταγιά να σας πει και θέλει να κάνει κάτι μέσω αυτού του νομοθετήματος για τις ΜΜΕ θεωρεί ότι έτσι θα διευκολύνει αυτούς που θέλουν να καινοτομήσουν, να εξαγάγουν να, να ε, ε, κινηθούν δηλαδή τις ΜΜΕ. Βεβαίω έχουμε εδώ και άλλου φραγμού και άλλα προβλήματα τα οποία θα μπορούσα να σα αναφέρω. Το διοικητικό άρθρο, το πρόβλημα στη ρευστότητα, τι δυσκολίε προσβασιμότητα στην, ε, στη δανειοδότηση, το ότι δεν μπορούν να προβληθούν στι αγορέ, ούτω ώστε να μπορούν να ψάξουν για επενδυτέ. Όλα αυτά είναι η τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, γιατί θα έχουμε εδώ μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων σχετικά τη ΜΜΕ και την αγορά εργασία. Οπότε και σε εκείνη τη μελέτη αναφέρθηκε ότι 3 εκατομμύρια θέσει απασχόληση τη ΜΜΕ κοστίζει αυτή η κρίση. Να γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση και δεν μιλούμε για κάτι νέο. Γιατί όλα αυτά μας έχουν απασχολήσει από το 2008, από τότε που είχαμε αυτή την εγκάρσια, την οριζόντια προσέγγιση που θα ήταν προσαρμοσμένη στι ανάγκες των ΜΜΕ και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, τελικά κατέληξε σε αυτήν την Small Business Act, αυτό το νομοθέτημα ε, για να μπορέσουμε να έχουμε απτή πρόοδο και να σας αναφέρω απλώς ε, το, το κόστος, το διοικητικό το οποίο θα πρέπει να συρρυκνωθεί έχουμε και άλλες ε, οδηγίες όπως είναι οδηγία για ε, την υπερημερία επίσης όσον αφορά και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ επίσης μας είπατε και εσείς κύριε Τρόιερ για τις ΜΜΕ ε, αυτό το τεστ το, οποίο ισχύει από το 2009 αυτό το οποίο ισχύει επί τη βάση ε, αυτών των προτάσεων και πρόσφατα σε μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, φάνηκε το τι απήχηση έχουν αυτά μας τα μέτρα της ΜΜΕ ε, και επίσης η οδηγία για την υπερημερία και όσον αφορά το πακέτο για την ομαλοποίηση νομίζω κύριε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο όπως και εσείς είπατε να ακολουθήσουμε την πρωτοβουλία του κ. Ταγιάννη και να έχουμε ένα εργαστήρι σε κάθε κράτο μέλος για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το τεστ των ΜΜΕ όσο γίνεται περισσότερο τον Φεβρουάριο. Επομένω, είχαμε αυτήν την Small Business Act, οπότε και εμεί δεσμευθήκαμε να αναβαθμίσουμε αυτό το τεστ και ο πρόεδρο Μπαρόσο τον ε, Ιούνιο είπε δύο λόγια στο Συμβούλιο όσον αφορά το τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, κυρίως όσον αφορά να δούμε τι θα κάνουμε με τις μικροεπιχειρήσεις, επίσης πώς θα προβληθεί προωθηθεί περισσότερο το τεστ αυτό και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Επομένως όλα αυτά ε, αποτελούν ένα, ένα μέσο πολιτικής πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς με την πολιτική μας για τις ΜΜΕ και θα πρέπει αυτό να ε, συμπληρωθεί όμως και με άλλα μέτρα τα οποία θα σας αναφέρω. Πρώτη προτεραιότητα είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατεβάσει ένα προπολογισμό 2,7 δις ευρώ για να τις υποστηρίξει τις ΜΜΕ και ελπίζουμε ότι στις επόμενες δημοσιογικές προοπτικές θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τις ε, υποστήριξη του Κοινοβουλίου και όσον αφορά τις συζητήσεις για τις επόμενες ε, τέτοιες ε, προοπτικές θα διπλασιάσουμε την πρεκοδότηση για τις ΜΜΕ ε και οπότε θα προσέξουμε τόσο ώστε αυτοί οι πόροι κατά προτεραιότητα να διατεθούν τις ΜΜΕ κατά την αρχική φράση φάση συγγνώμη, της ανάπτυξής τους που είναι η πιο σημαντική φάση και εκεί είναι οι πιο ευάλωτες αυτές οι ΜΜΕ. Επίσης αυτή η πρικοδότηση θα ωφελήσει και όσον αφορά να δούμε πώς θα έχουν καλύτερη προσβασιμότητα σε χρηματοδότηση δράσεις στον πρώτο κεφάλαιο παιχνικού κινδύνου όσον αφορά το χρηματιστήριο και όσον αφορά την τραπεζική πίστη. Όλα αυτά τα ξέρετε όσον αφορά ε, ότι εγώ τα έχω αναλάβει αυτά στο προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο και όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όλα αυτά θα τα καλύψουμε με το Single Market Act ε, και θα μπορέσουμε αυτή την, ε, την, τη κάνουμε μια εκδήλωση να κάνουμε κάποια μέτρα για να βοηθήσουμε τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην Ευρώπη ούτω ώστε να καταλήξουμε ή στο να έχουμε ένα, ένα ταμείο capital risk ε, επαγγελματικού κινδύνου. Εγώ σε συνεργασία με τον κύριο Ταγιάννη θα το προωθήσουμε αυτό και να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με τα με κατόφλια τα οποία εμποδίζουν πάρα πολλέ ε, ΜΜΕ να μπουν στο χρηματιστήριο και επίση πώ θα βελτιώσουμε την πάρα πολύ περιορισμένη ε, ε ρευστότητα. Κύριε Τζαβέλα, μα αναφέρεται και κάτι άλλο. Μα αναφέρεται και τα τη τραπεζική πίστη και την προσβασιμότητα. το πρόβλημα αυτό είναι το πρόβλημα τη κρίση. Ότι τώρα λοιπόν έχουν κλείσει οι αυτό θα πρέπει να το δούμε τις τράπεζες και θα πρέπει επίσης να προσέξουμε κύριοι βουλευτές γιατί η νομοθεσία αυτή την οποία προπαρασκευάζουμε και σας είπα και τον Ιούλιο από τη βάση των, κανόνων της Βασιλείας από τη βάση της ρευστότητας, της χρηστής ε, διαχείρισης ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται και ε, επί των ΜΜΕ ενώ ήδη έχουμε 8.300 τράπεζες ξέρετε που αυτές χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία οπότε ήδη έχετε κάποια μέτρα στην πατρίδα σας σε σχέση με αυτά επίσης κάτι άλλο πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τις ΜΜΕ είναι το ότι αποτελούν το, το, την, την καινοτομία και ε, θα μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε την έρευνα και τεχνολογία στο, στα πλαίσια της πολιτικής μας με τον ΕΣΤΟ 2020, ε, έρευνα επίση ε, συμμετοχή στον, ε, στον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, να δούμε πώς επομένως για με το 2012 να, να τις βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να χρηματοδοτηθούν αυτές που ασχολούνται με καινοτομία και έρευνα οπότε έτσι να, να αποκτήσουν αυτή την πρικοδότηση που προβλέπουν των 120 εκατομμύριων ευρώ και επίσης να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των ΜΜΕ εις τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης των ε, διορθωτικών ταμείων. Ναι, και εγώ και άλλοι αδελφοί μου θέλουμε να μπορούν να έχουν περισσότερη προσβασιμότητα ΜΜΕ σε αυτό το ταμείο. Θέλουμε με τον κανονισμό των ε, διορθωτικών ταμείων να τις βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Μεγάλη μας επίσης προτεραιότητα είναι το πώ θα έχουμε λιγότερη δικαιωτική γραφειοκρατία τη ΜΜΕ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δράση. Ε, θα το προωθήσουμε φέτος, του χρόνου μάλλον, συγγνώμη, του 2012 και πάμε για μείωση κατά ένα τέταρτο αυτής της ε, διοικητικής ε, των διοικητικών υποχρεώσεων της γραφειοκρατίας και να δούμε τι θα γίνει με τη λογιστική των μικρών επιχειρήσεων και αυτές οι προτάσεις θα υιοθετηθούν τάχιστα, έχουμε 120 προτάσεις συνολικά για να μειώσουμε μέχρι και 31% τη γραφειοκρατία, τη διοικητική, οπότε πάμε για μείωση 22% των σχετικών τελών που επιβάλλει η διοίκηση. Άλλη μας προτεραιότητα είναι το ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε την καινούργια μας συνεκτική στρατηγική για να μπορέσουμε να διευκολυνθεί η προβασιμότητα των ΜΜΕ στις ε, δημόσιες συμβάσεις ε, και γι' αυτό και θα προσθέσουμε τις, ε, τους διαγωνισμούς τις συμβάσεις γι' αυτό το έχουμε πει, το έχουμε εξαγγείλει και προσωπικά και όλη η Επιτροπή και γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει καλή προσβασιμότητα στις διεθνείς αγορές και πώς θα μεταφερθεί η συμφωνία GPA εις το κοινωτικό δίκαιο και τελικά να έχουμε κάποιε αγορές που να μπορούν να τις ε, εκμεταλλευτούν και θέλουμε να υπάρχει ομαλοποίηση ε, και αυτό θα γίνει με την προσαρμογή της νομοθεσία τα ΜΜΕ. Θέλουμε επομένως να υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ όλων όσων ασχολούνται. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια ιδεολογήματα φορτισμένη νομοθεσία δηλαδή με ιδεολογήματα. Θέλουμε επομένω έτσι να προχωρήσουμε γιατί κάνετε συγκεκριμένε ερωτήσεις με το Single Market Act γιατί έχουμε αυτά τα 12 επιμέρου ε, μέτρα τα είπαν ε, όλοι οι συνάδελφοι και έχουμε τις 50 ε, προτάσεις για αυτά τα 12 σημεία κλειδιά πρόκειται για νομοθεσία η οποία είναι νομοθεσία πρωτοβουλίας, νομοθεσία που διευκολύνει το έργο των ΜΜΕ. Να, επομένως, αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα. Να, είναι και το, Ευρωπαϊκό Μαύρες Τεχνία που εσάς σα ενδιαφέρει. Και ακριβώς λόγω ε, της ε, τιμής του είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούν να έχουν προσβασιμότητα οι ΜΜΕ. Να, όλα αυτά για τι ΜΜΕ και ο κύριος Κρέσπος σας τα είπε, ε, κάποιο τρόπο έγινε ο πρέσβης των ΜΜΕ. Στις 14 Σεπτεμβρίου έγινε μια εκδήλωση που ακριβώς αφορούσε αυτό το θέμα. Το πώς θα έχουν πρόσβαση στην ε, πίστη, στα δάνεια, η ΜΜΕ. Αυτό βέβαια θα γίνει με όλε τι ελληνικέ αρχέ, οι οποίες είναι οι υπεύθυνε τόσο ώστε να εφαρμόσουν αυτή μας την νομοθεσία, το σύγκλημα αρκετά και όλε μας τι πρωτοβουλίες για τις ΜΜΕ, ούτω ώστε οι επιχειρήσει οι ευρωπαϊκές να αντιμετωπίσουν την κρίση και έτσι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ε, ανταγωνιστικότητας και έτσι θα πρέπει γι' αυτό να τις βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ Επίτροπε Μπαρνιέ και τώρα εξ ονόματος των ομάδων ε, ο κύριος Μπένσεν 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Επίτροπο γιατί πραγματικά ανέλαβε δέσμευση υπέρ των ε, ΜΜΕ. Αυτή η νομοθεσία είναι η ομπρέλα που πρέπει να καλύπτει την νομοθεσία για το θέμα αυτό. Τρία θέματα είναι σημαντικά εδώ. Η πρόσβαση στα κεφάλαια είναι το πρώτο, δεύτερον πρόσβαση στις αγορές, και αυτό το συζητήσαμε, και τρίτον μείωση του διοικητικού φόρτου. Σίγουρα η οικονομική ύφεση δυσκολεύει πάρα πολύ τις ΜΜΕ ως προς την πρόσβαση σε κεφάλαια. Και περιμένω τώρα την πρόταση της Κομισιόν που θα ε, εγγυάται ότι θα είναι υγιείς, λειτουργικές, ΜΜΕ και θα έχουν και πρόσβαση σε κεφάλαια. Τώρα για την πρόσβαση στις αγορές, βέβαια για αυτό το πράγμα πρέπει να λειτουργεί καλά η εσωτερική αγορά και η ΜΜΕ πρέπει να συμμετέχουν στο εμπόριο με την Κίνα κλπ αν θέλουμε να αυξήσουμε και εμείς όπως εκείνη το ποσοστό με την με ανάπτυξη πρέπει να έχουμε διασφαλισμένη την πρόσβαση στις αγορές τους. Και πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας είναι πολύ σημαντική. Και τα εθνικά κράτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να νοικοκυρέψουν τα του οίκου τους για αυτό το πράγμα αν πρόκειται να εφαρμόσουν την οδηγία η οποία θα διασφαλίσει βέβαια κεφαλαϊκή επάρκεια στις τράπεζες με πρόβλημα ε, συνεπαγόμενο ίσως για τις ε, ε μημία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόγια. Ευχαριστώ. Η ευρωπαϊκή κρίση μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο μεταξύ όσον αφορά την συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει ύφεση. Εάν λοιπόν δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα της ΜΜΕ θα ήθελα η Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη αυτές τις αρχές και να υπάρξουν ε, πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου όπως το Small Business Act με αποτελεσματικότητα και ποιότητα γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις πληρωμές. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΜΜΕ. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε κατά πόσο όταν νομοθετούμε το κάνουμε υπέρ των ΜΜΕ. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και να δημιουργήσουμε αυτή την πλαισίωση, όπως είπατε, γιατί εκτιμούμε και την εργασία της Κομισιόν και θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες διαγράφονται. Κύριε Επίτροπε, ας είμαστε σαφείς ως προς τράπεζες γιατί θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Κόβει τον λόγο. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε κύριος Βάτσον τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαιρετίζω την πρώτη, τις προτάσεις της Κομισιόν και χαιρετίζω και το έργο της εισηγήτριας των, των εισηγήσεών μας. Ε, οι ΜΜΕ δημιουργούν απασχόληση, είναι οι κινητήριες δυνάμεις μας, είναι τα έμβρια των μεγάλων επιχειρήσεων. Κατά το παρελθόν παραγνωρίστηκαν συχνά από τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τους μεγάλους εργοδότες και τη βιομηχανία. Κλειδί για την επιτυχία τους είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδότησης ήταν πολύ σημαντικό και στη δική μου περιφέρεια και χαιρετίζω τη δέσμευση του Επιτρόπου να εξετάσει νέες ευκαιρίες για το κεφάλαιο το επιχειρησιακό. Επιτρέπεται ενδιάμεση ερώτηση, εμβόλυμη από τον συνάδελφο Μάρτιν. Ο κύριος Μάρτιν, δεν ήθελα να διακόψω, ήθελα να ακούσω τι θα πείτε και μετά θα έθετα την ερώτηση. να περιμένει και να με ρωτήσει μετά. Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το, το σύστημα το τραπεζικό όταν επανακεφαλαιοποιηθεί θα δανείζει πάλι στις μικρές επιχειρήσεις. Χαιρετίζουμε ε, τις προτάσεις για τις καθυστερημένες πληρωμές από την Κομισιόν. Πρέπει να κάνει κάτι για να απλουστεύσει και το ΦΠΑ ιδιαίτερα στις διασυνοριακές συναλλαγές. Εγώ πήγα στο Φάντραξ, στο Σάμαρτον, στην εκλογική μου επιφέρεια και μου λένε ότι 27 κατόφλια ΦΠΑ λειτουργούν αυτή τη στιγμή και δυσκολεύονται πολύ να εμπορεύονται οι μικρές επιχειρήσεις. Ελπίζω να δει και τον νόμο για την απασχόληση κομισιών που προβλέπει εκτιμήσεις επιπτώσεων και καμιά φορά και ρήτρε τερματισμού σαν σέτη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν τώρα την εμβόλυμη. Κύριε Βότσον, είστε έμπειρος βουλευτής και γνωρίζετε τα θέματα αυτά ποιες πρόοδοι έγιναν ε, όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των ΜΜΕ. Βλέπετε πρόοδοι ή μήπω είμαστε στα ίδια και στην υπερβολική γραφειοκρατία. Ξέρετε την Κίνα. Θα λέγατε ότι η ΜΜΕ στην Κίνα υπόκεινται σε λιγότερες ρυθμίσεις από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βάτσον, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι για την ερώτηση. Πράγματι εργάστηκα και στην ε, ε, Κίνα και είδα τις δυσκολίες που υπάρχουν και εκεί για τις ΜΜΕ. Οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές, αντιμετωπίζουν όμως πολλές προκλήσεις που δεν έχουν οι δικές μας. Ε, το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ ελπίζω να έχει τώρα κατατεθεί και ελπίζω η Κομισιόν να δώσει βάση σε θέματα φθηνότερη ενέργεια, ε, ευρύ, τεχνολογίες ευρέως φάσματος, ώστε να βοηθηθούν και να αναπτυχθούν και να ευημερίσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ με τον Επίτροπο γιατί στη Βόρεια Ιρλανδία το 99% των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ στην εκλογική μου περιφέρεια. Εξαρτώμεθα για την ανάπτυξη σε αυτές και η, τώρα ο αντίκτυπος στην περιφερειακή οικονομία λόγω της κρίσης είναι ε, μεγάλος. Όλες δουλεύουν ε, κατά από σκληρές συνθήκες, αντιμετωπίζουν πολλές πιέσεις και βεβαίως ε, το θέμα το, της δανειοδότησης είναι σημαντικό και τεράστιο πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα είναι η γραφειοκρατία που πρέπει να καταπολεμούν και να αντιπαρέρχονται σε καθημερινή βάση. Άκουσα με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Επιτρόπου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για τις μικρές επιχειρήσεις και αυτό το τεστ των ΜΜΕ ώστε να αναλυθεί η νομοθετική επίπτωση στο, στις μημία στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην Ευρώπη όμως να μην υπεριθμίσουμε την αγορά γιατί τότε ε, άλλοι θα ε, αναπτυχθούν σε βάρος μας. Ευχαριστώ ο κυρίος Beauty Coffer. Τρία λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η νομοθεσία για τις ΜΜΕ είναι καλό νομοθέτημα, αλλά δεν είναι νόμος, ε, είναι μια διακήρυξη. Αν θέλουμε η Κομισιόν, όπως είπε ο κύριος Στόιρ, να δράσει υποδειγματικά για τις ΜΜΕ, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα δύο σημεία. Τα θέματα ε, που αφορούν τα χρήματα και τα θέματα που αφορούν τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Θα πω δύο πράγματα εδώ. Καταρχήν το πρόγραμμα έρευνας. Δεν είμαι, εξακολουθώ να μην είμαι ικανοποιημένο. Έχουμε τη Γενική Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις, έχουμε τη Γενική Διεύθυνση ε, έρευνα και έκαναν διαπραγματεύσεις για το μέλλον αυτού που λέγαμε πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία το οποίο είναι ευνοϊκό, θετικό για τις ΜΜΕ, φιλικό για αυτές. Όμως η επιχειρηματική επιχειρηματικότητα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον. Πάντως ένα θα πρέπει να είναι το κριτήριο του Κοινοβουλίου προς την Κομισιόν για τις ΜΜΕ. Δεν ε, τις ενδιαφέρει μόνο η χρηματοδότηση αλλά και η ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα, πιο εύκολη από ό,τι μέχρι τώρα. Και βέβαια είναι ευρεία η έννοια των καινοτομιών. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα όταν οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ πριν από λίγες εβδομάδες ε, ήρθαν στις ε, Βρυξέλλες για τη βδομάδα των ΜΜΕ και ένα βασικό θέμα το οποίο μας επεσήμαναν είναι ότι η καινοτομία δεν περιλαμβάνει μόνο την έρευνα. Ιδιαίτερα το λέω για τις ΜΜΕ και η καινοτομία των ΜΜΕ μπορεί επίσης να συμβάλλει στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να τους διασφαλίσουμε ακόμα καλύτερη πρόσβαση και να μην τις εξαρτούμε από τις ε, ε, μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη έρευνα. Εδώ πρέπει να δείξει η Κομισιόν ότι αυτό το οποίο διακηρύσει Θεωρητικός μπορεί και να το εφαρμόσει υπέρ των ΜΜΕ. Δεύτερον, διαρθρωτικά ταμεία. Ο κύριος Μπαρνιέ το ανέφερε αυτό ευτυχώς. Εκεί η πρόσβαση για τις ΜΜΕ πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Θα πρέπει να υπάρξουν τοπικές εταιρικές σχέσεις, περιφερειακές μεταξύ δημοσίου, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ΜΜΕ. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα. Ε, υπάρχουν ε, κάποια innovation vouchers ή το Steinbytes ή το Cambridge που μπορούμε να, από εκεί να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Επίσης, τις κυβερνητικές ε, δομές θα πρέπει να εντάσσονται περισσότερο, να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες. Είναι κρίμα που η Κομισιόν δεν κατάφερε στην πρόταση για την ανανέωση της τυποποίησης να εντάξει περισσότερο της ΜΜΕ και να τους δώσει δικαίωμα ψήφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιτικόφερ. Ο κύριος Προβέρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αναφέρομαι στον τομέα που γνωρίζω καλύτερα, τη Βόρειο Ιταλία. Και το πιο σημαντικό για τις ε, ΜΜΕ είναι η δανειοληψία. Αυτό μας απασχολεί πολύ περισσότερα από τη γραφειοκρατία, το διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από πλευράς ε, Κίνας οι τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιώσουν, κεφαλαιοποιήσουν με συγχωρείτε, και δεν δίνουν, δεν χορηγούν δάνεια στις μικρές επιχειρήσεις γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες εγγύησεις. Γι' αυτό, παρά την καλή τους θέληση, δεν προχωράει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί δανειοδότησης που θα βοηθούν ως προς την, τις ε, πληροφορίες που χρειάζονται γιατί χωρίς χρήματα δεν υπάρχει έρευνα, δεν υπάρχει δυνατότητα επενδύσεων και άρα δεν μπορούμε να προωθήσουμε την ευημερία μιας χώρας. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Όλοι το ξέρουμε και όλα τα έχουμε πει Εγώ όμως θα σας επενέσω κύριε Επίτροπε. Αυτά που είπατε είναι σημαντικά, σωστά, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η πραγματικότητα όταν ε, έχει κανείς να κάνει με εκπροσώπους των ΜΜΕ ε, δείχνει ότι ακόμη απέχει πολύ από αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως ό,τι αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Τα νούμερα τα ξέρετε, μόνο 34% όλων των δημοσίων διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν στις ε, ΜΜΕ παρόλο που ε, ως προς την οικονομική τους παραγωγικότητα ε, αποτελούν το 50%. Υπάρχει λόγος, ε, έχει να κάνει με την συγκεκριμένη τους δραστηριότητα. Ε, είναι μεγάλες οι πιέσεις. Βέβαια, καλό είναι να είμαστε αισιόδοξοι και παλιά είχα την ευκαιρία να κάνω εκθέσεις στην, Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή ε, όπου μιλήσαμε για ε, στατιστικές και πιο εύκολη πρόσβαση, αλλά σε τελευταία ανάλυση το πρόβλημα είναι η δυνατότητα κατανόησης όλων αυτών των δυνατοτήτων οι πύλες, ε, η πρόσβαση σε αυτές, πώς θα, χωρίς πολλή γραφειοκρατία, θα ε, μπορέσω να αποκτήσω κεφάλαια, να έχω πρόσβαση σε αυτά. Σε αυτό το θέμα νομίζω ότι θα έπρεπε να αφιερώσετε περισσότερη προσοχή. Ευχαριστώ, κυρία Ντελκαστίγιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, Έχουμε σταθεί ή τα θέματα τα χρηματοπιστωτικά για την ρευστότητα, για τις τραπεζικές πιστώσεις, τη δυσκολία προσβασιμότητας. Ε, είναι συμβαρό αυτό όρομος, αυτό είναι πρόβλημα των ΜΜΕ, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων, των τραπεζών, αλλά πάνω απ' όλα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό είναι πρόβλημα όλων, όλων, καθενός, καθεμιάς από τους πολίτες του Ευρωπαίου, Εγώ θα ήθελα τώρα να σταθώ σε μια διάσταση που φαίνεται πάρα πολύ σημαντική και είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ ελαφρά το θίξαμε. Είναι κάτι το οποίο αφορά την εσωτερική αγορά. Διότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε εδώ πέρα σταθεί στα θεσμικά όργανα το πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε κάτι αποφασιστικό για να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά. Θεωρούμε ότι είναι στρατηγικός παράγοντα για να βρούμε το διέξοδο, τι το διέξοδο από την κρίση. Και αν κάτσουμε να δούμε ποια είναι η σχέση με εξωτερική αγορά και τον ΜΜΕ, θα διαπιστώσουμε ότι μόνο το 23% των ΜΜΕ έχουν διασυνοριακέ συναλλαγέ και μόνο το 13% το κάνει πέρα από τα σύνορα της, του, του, του κράτους. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτό το τεράστιο χάσμα των ε, ελλημάτων. Άρα θα πάμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την κατάτμιση της νομοθεσίας που μας οδηγεί στο πρόβλημα της ε, εσωτερικής αγοράς. Τι γίνεται όσον αφορά τη σχέση κόστος αποτελέσματος. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο επομένως να κάτσουμε και να χρηματοδοτήσουμε, να υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά αυτή την, την κατάτμιση της κοινωτικής νομοθεσίας σε σχέση με τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Τελικαστήγιο. Τώρα η κυρία Μέρκες για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Αυτό το οποίο τώρα λέμε είναι το τι θα κάνουμε στην σημερινή συγκυρία της κρίσης και λέμε θα πρέπει να προσέξουμε το τι θα κάνουμε με τις ΜΜΕ. Δεν μιλάμε όμως μόνο για το χρήμα που είναι σημαντικός παράγων. Που θέλω να δούμε είναι να βρούμε τι γίνεται όσον αφορά την κατάλληλη ε, εκπαίδευση. Ε, δηλαδή να δούμε πώς η καινοτομία θα υπάρχει, θα χρησιμοποιείται όμως επίσης. Πάρα πολλοί μιλούν για έρευνα, όμως δεν μιλούμε αρκετά για καινοτομία και για μία Νομίζω θα πρέπει να κάτσουμε και να επικεντρωθούμε περισσότερο ή στα χρηματοοικονομικά ή στο χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό σύστημα διότι πάρα πολλοί κάθονται και μας μιλούν για κάποια μικρά ποσά τα οποία χρειάζονται ε, το, το μάνα εξ ουρανού, το, το κεφάλαιο, τη χρηματοδότηση, μα πώς θα γίνει αυτό το ταμείο που θέλει να φτιάξετε, θα τα καλύψει όλα, θα καλύψει και τα μικρά ποσά ε, γιατί πάρα πολύ συχνά έρχονται κάποιοι, κάποιες επιχειρήσεις πάνε να κάνουν μια δεύτερη αρχή. Μα χρειάζεται να του δοθεί μια ευκαιρία. Και ο κύριο Σταγιάννη έρχεται και μα λέει ότι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Κομισιόν, δεν είναι τόσο καλή όσον αφορά το να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στι επιχειρήσει. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, μπα και μπορούμε να βελτιώσουμε το, το σχετικό θέμα, να δούμε πώ θα μπορεί ο κόσμο να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Ε, ένα λεπτό, κύριος Γκάλαχαρ. Ευχαριστώ. Η, στην Ιρλανδία 250.000 ε, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, υπάρχουν για την ε, απασχόληση. Είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα όμως η πρόσβαση ε, στο, στη χρηματοδότηση. Ε, σήμερα πολλές ζωτικές επιχειρήσεις ε, παλεύουν να αντιμετωπίσουν την ύφεση. Και βέβαια το θέμα της απειλής των θέσεων εργασίας είναι πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος Μπαρόζο έκανε μία, ε, ανέλαβε μία δέσμευση ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Το μέσο του ΜΜΕ είναι η κινητήρια δύναμη της βιομηχανίας της. Πρέπει να τις βοηθήσουμε με πολιτικές ε, που θα δημιουργούν θετικό οικονομικό κλίμα ευεπίφορο για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαχαρ. Και τώρα ο κύριος Στοσενόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αυτονόητο ότι όλοι θεωρούμε πολύ ζωτική σημασία το ρόλο των ΜΜΕ και νομίζω ότι θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και πόσο γνωρίζω από πολλούς επιχειρηματίες εκτιμούν αυτή την προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνούμε τους ε, κανόνες που έχουμε εισαγάγει και εγκρίνει, διότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα ΜΜΕ, μιλάμε για την υποχρεωτική σήμανση, ε, υποχρεώσεις προς εστιατόρια και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με μία ε, διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία που επιβαρύνει τις ΜΜΕ. Επίσης, όταν εισαγάγεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όταν μιλάμε για ε, προσωπικό το οποίο προσλαμβάνει μια επιχείρηση, θα πρέπει να ξέρουμε τι επιπτώσεις υπάρχουν. Ευχαριστούμε. Μοργάντη για μισή λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Έχει μεγάλη σημασία, έχουν μεγάλη σημασία οι ΜΜΕ για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαδικασία δανειοληψίας με βάση τη Βασιλεία 3. Και νομίζω ότι με βάση τους κανόνες της Βασιλείας 3 η διαδικασία αυτή θα είναι πιο δαπανηρή διότι προαπαιτεί ένα πολύ υψηλό κεφάλαιο έτσι ώστε να χορηγηθεί δάνειο και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και το κόστος της χρηματοδότησης που θα πλήξει τις ΜΜΕ. Εάν λάβουμε υπόψη ότι τα δάνεια αυτά δεν είναι υψηλού κινδύνου δεν θα μπορούσαμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να καινοτομήσουμε. Μπορούμε όμως να καινοτομήσουμε χωρίς τους κατάλληλους πόρους. Ευχαριστώ κύριε Μοργάντη. Ο κύριος Μπρόνς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. 10% των ΜΜΕ μόνο εξάγουν σε άλλα κράτη-μέλη και σε λιγότερες ακόμα χώρες εκτός Ευρώπης. Πολλές ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με πολύ λίγους εργαζομένους. Τα γραφεία ε, που παρέχουν, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ε, στην Κίνα δεν φτάνουν ε, στις μικρές αυτές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι μικρές λοιπόν, όταν ερωτώνται τι θέλουν από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία ή αυτή την εγγύηση ή αυτή την επιδότηση θέλουν απαλλαγή από υπερβολικές ρυθμίσεις και καταπιεστική φορολόγηση. Μέχρι το 2010, από το 2008 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 100, ε, ήταν, ήταν ε, πολλές χιλιάδες οι επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε άλλες υπήρους. Ε, ε, αναφέρομαι πολλά ε, τα οποία όμως τορπιλίζονται από το ευρωπαϊκό δόγμα. Ευχαριστώ κυρία Μπρόνς, η κυρία Σαρτόρη 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα για την ευρωπαϊκή οικονομία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν και διαστάθηκαν και ένιωσαν την ε, κρίση, τα κατάφεραν πολύ καλά και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από όλα τα στοιχεία που διάβασα, μπορώ να πω ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες έχουν έδρα στα κράτη-μέλη που είναι επικεφαλής ε, στους τομείς της ε, καινοτομίας ανακτούν το χαμένο έδαφος πολύ πιο εύκολα από άλλες χώρες που δεν παρουσιάζουν καινοτομίες. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος που ακολουθεί η Ευρώπη μέσω της στρατηγικής 2020 και ο ρόλος που προσδίδει στην καινοτομία είναι και ο σωστός. Θα πρέπει όμως να αποδώσει τάχιστα πολύ πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε και είχαμε εξαγγείλει το 2009. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και θα πρέπει να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες. Από την παρέμβαση του, Επιτρή, του Επιτρόπου άκουσα πολύ σημαντικά αριθμητικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία ένα έκρινα άκρος ενδιαφέρον το ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις μικροεπιχειρήσεις και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δράσουν πιο εύκολα. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρτόρη. Ο κύριος Κούτας έχει το λεπτό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η χρηματοοικονομική ε, κρίση έχει πλήξει τις μικρομεσές επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τις καινοτομίες. Το 55% των ΜΜΕ το 2010 έδειξαν χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με το 2009. Ε, αν λάβουμε υπόψη τη σημασία των ε, δραστηριοτήτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την αγορά εργασίας και αν λάβουμε υπόψη ότι το 67% των θέσεων εργασίας προέρχονται από ΜΜΕ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, θα, ότι οφείλουμε να τις ενθαρρύνουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να άρουμε τα γραφειοκρατικά προσκόμματα. Κάνουμε πολλές επενδύσεις για να σώσουμε το τραπεζικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι εξίσου σοβαρές προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλουμε για να σώσουμε τις μικρομεσαίες. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ε, το λόγο έχει ο κύριος Ρινάλτη. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι αν ακούγαμε τη φωνή ενός μικρού επιχειρηματία θα ακούγαμε μια φωνή γεμάτη ανησυχία. Ιδιαίτερα ως προς τα διαρθρωτικά προβλήματα που γνωρίζει αυτός ο τομέας. Δηλαδή, χρειάζεται βοήθεια για τη διεθνοποίηση. Μιλάμε για την άρση της γραφειοκρατίας, γιατί μόνο για την καταβολή του ΦΥΠΙΑ υπάρχει, εν υπάρχει μεγάλο κόστος. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σωστή και επαρκής πρόσβαση στα δάνεια. Δεν έχει νόημα ε, να αναδιαρθρώσουμε τις τράπεζες εάν δεν υπάρχει πίστη προς ένα τομέα ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες μας όπως η ΜΜΕ. Ε, σήμερα τις εκβιάζουμε και τις εξουθενώνουμε. Αυτό γίνεται τουλάχιστον από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό ο κύριος ε, Πάσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι παρά το ότι έχουμε εκτεταμένη παρέμβαση των θεσμικών οργάνων, όσον αφορά τις ΜΜΕ, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα του νομοθετικού ε, περιβάλλοντος, διότι σύμφωνα με τις, ΜΜΕ δεν προσέχει η διοίκηση. Ε, υπάρχουν θέματα και όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και θα πρέπει κατά τη δική μας άποψη να προσπαθήσουμε να άρουμε τους φραγμούς που είναι η γραφειοκρατία, το διοικητικό βάρος και στη δική μας χώρα. Θα πρέπει ένα σωρό έντυπα να υποβάλλονται σε ένα σωρό αρχές και επομένως θα πρέπει να μειωθεί αυτό. Θα πρέπει λοιπόν στις χώρες αυτές ε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται στην Κίνα, τι γίνεται στην Ινδία. Είναι οι ανταγωνιστές μας. Αυτοί κάνουν δουλειά τους και πληρώνουν και φόρους. Ε, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ε, το πόσο σκληρή είναι η κρίση ιδιαίτερα στις, ε, για τις ΜΜΕ. Ε, στραγγαλίζονται κυριολεκτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια μελέτη για τις ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές αγορές και ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει τη στρατηγική, τη της, αλλά τα βασικά προβλήματα δεν λύνονται. Γιατί οι γραφειοκρατικές ελαφρύνσεις που τους υποσχέθηκαν δεν λειτουργούν. Το 99% των ε, ε ΜΜΕ ε, είναι μικρές. Παρόλα αυτά όμως αποτελούν ένα μεγάλο εργοδότη και είναι σημαντικό να τις προστατέψουμε απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να μπορέσουν να υποστηριχθούν γρήγορα και με ευέλικτο και αντιγραφειοκρατικό τρόπο. Ε, ο κύριος Ρούμπι είχε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μπαρνιέ. Νομίζω ότι το σημαντικότερο το είπε ο Υπουργό Οικονομικό της Τσεχίας Μίκλος τη Σλοβακία Μίκλος, που είπε ότι ε, η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό αναλαμβάνοντας και κάποιο ρίσκο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, τα προϊόντα, της, ε, ε, τη ρευστότητα που θα πρέπει να υποστηριχθεί ε, γιατί έτσι συνεχίζουν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες και δημιουργούν εμπιστοσύνη στην αγορά. Πάνω σε αυτή τη βάση θα ξαναγίνει η ανταγωνιστική Ευρώπη. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις μας να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και γι' αυτό χρειάζεται μια στρατηγική εκπαίδευση και επιμόρφωσης είναι ε, πολύ σημαντικό να ανανεώσουμε το εργατικό μας δυναμικό και το ειδικευμένο δυναμικό αρχιτέκτονες ε, κλπ. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ελέγξουν το θέμα της φορολογίας των επιχειρήσεων και να δουν αν είναι σωστή. Η Βουλγαρία έχει 10% φορολόγηση κερδών. Η Ελλάδα από την άλλη έχει την υψηλότερη 40% φορολογία επί των κερδών και προφανώς οι επιχειρηματίες αρνούνται να πληρώσουν τόσο υψηλό φόρο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε μαθήματα ε, από αυτή την κατάσταση και να καταλήξουμε σε μια, ένα βέλτιστο ποσοστό ε, φορολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρινς για μισή λεπτό. Πρόεδρε. Όλοι μιλούμε για την κρίση. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όμως θα πρέπει να μας απασχολήσουν όχι μόνο τα αίτια της κρίσης, ο τραπεζικός τομέας, το ε, δημόσιο χρέος, αλλά ποια είναι η οδός διαφυγής. Αυτό θα το καταφέρουμε όταν ε, βρεθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Όμως αυτές οι νέες θέσεις απασχόλησης δεν θα δημιουργηθούν στον τραπεζικό τομέα ούτε από τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά από τις μικρές και μεσές που απασχολούν 90 εκατομμύρια ανθρώπους ανά την Ευρώπη. Για να υπερβούμε την κρίση λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις ΜΜΕ οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα και μπορούν να διδαχθούν από τα σφάλματά τους. Επίσης, μπορούν να δράσουν άμεσα για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των αγορών και επίσης μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή να προσλάβουν ε, νέους ανθρώπους. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να βοηθήσουμε αυτό το τομέα. Καταρχήν να κρατήσουμε τα σύνορά μας ανοιχτά να δώσουμε χρηματοοικονομικές ευκαιρίες μέσω venture capital και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία που αποτελεί πρόσκομα στην ανάπτυξη. Η ΜΜΕ θα μας βγάλουν από την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό και ο συνάδελφος Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό το θέμα απόψε και ε, δεδομένων των ε, γενικότερων συνομιλιών. 22,5 ε, εκατομμύρια άνεργοι, 23 εκατομμύρια ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να το συσχετίσουμε αυτό σε σχέση με την ασφάλεια της απασχόλησης στην Ευρώπη κάτω από τις ε, θετικές ε, και τις σωστές συνθήκες θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και βεβαίως ε, μια προϋπόθεση είναι η χρηματοδότηση. Όταν κεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες στη χώρα μου, δυσκολεύτηκαν οι όροι προς τις ΜΜΕ ε, αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν ε, παρήχαν σχεδόν καμία διευκόλυνση. Επίσης, ο Επίτροπος μίλησε για την ανάγκη απλούστερης ρύθμισης για τις ΜΜΕ σε ό,τι αφορά δημοσίες συμβάσεις κλπ. Και μίλησε και για τη σημασία του κεφαλαίου κινδύνου. Εμείς ε, θέλουμε να το με το κεφάλαιο κινδύνου να υπάρχει, γιατί είμαστε πίσω τουλάχιστον σε σχέση με τις ΗΠΑ γιατί ε, έτσι θα δημιουργηθούν καινοτομίε. Τώρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχουν διάφορες στατιστικές. Ε, εδώ σίγουρα ανοίγεται θαυμάσια ευκαιρία να βοηθηθεί και η οικονομία και η μημία και η απασχόληση. Ευχαριστώ συνάδελφε Κέλλη. Πάμε στη διαδικασία Catch the Eye και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Σουάμπ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πολλά είπαμε για τις ΜΜΕ. Ε, οι κανόνες για αυτές πρέπει να ισχύουν ε, όπως και για όλους. Εμείς δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες ε, μετά την δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Οι ΜΜΕ θέλουν ένα περιθώριο κίνησης ε, το οποίο δεν έχουν ε, την πρόσβαση σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και με ε, άλλες οδηγίες να βοηθήσουμε και να εναρμονίσουμε το νομοθετικό καθεστώς στην Ευρώπη ώστε με ενιαία πρότυπα να καλύπτεται η αγορά. Ε, θέλουμε τέτοια παραδείγματα και σε άλλους τομείς γιατί οι ΜΜΕ δεν έχουν εξειδικευμένο ενδιαφέρον, θέλουν μόνο ε, ενιαίους και εναρμονισμένους κανόνες. Και πάνω σε αυτό πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Χάντσλικ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, είμαι σκιώδης ε, εισηγήτρια για την οδηγία των καθυστερημένων πληρωμών και υπάρχουν πολλές ανισορροπίες σε σχέση με την κατάσταση των ΜΜΕ στα διάφορα Δηλαδή δεν υπάρχει ισόβαθμη μεταχείριση. Πολλές φορές η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ε, δυσχερής και επιδεινώθηκε η κατάσταση των ΜΜΕ, ιδιαίτερα αν δούμε με ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Βλέπουμε ότι μόνο για λίγες ε, μικρές επιχειρήσεις έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χαίρομαι διότι θα κάνετε έκκληση προς τον ε, Επίτροπο Ταγιάννη για να εκτελέσει αυτή την οδηγία, να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η οδηγία για τις ε, καθυστερημένες ε, πληρωμές. Ευχαριστώ κυρία Χάνσλικ. Η κυρία Μπασέσκου. Καταρχήν, οι ΜΜΕ συμμετέχουν όσο καλύτερα μπορούν σε αυτό το πλαίσιο. Το Small Business Act που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008 προωθεί τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις έτσι ώστε να παγιώσει την ανταγωνιστικότητα. Έχει σημασία η κατάρτιση και η εκπαίδευση ως προς τις ε, βέλτιστες πρακτικές και στη χώρα μου το πρόγραμμα START δίνει νέες ευκαιρίες στους ε, νέους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ΜΜΕ για να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και επίσης να δημοσιοποιείται το έργο τους. Έτσι μπορέσαμε να σώσουμε 300.000 θέσεις εργασίας. Επίσης η Ρουμανία προώθησε την χρηματοδότηση του ΜΜΕ μέσα από ένα δημόσιο πρόγραμμα πολιετούς διάρκειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λούχαν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2008 εγκρίθηκε το Small Business Act και βοήθησε τις μικρές επιχειρήσεις, όμως ε, θα ήθελα αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης να, να τεθεί υπόψη, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς δρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια της ε, ε, του δραστηριότητα, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξοικονομήσουμε χρόνο και βοήθεια μέσω αυτού του πλαισίου ε, νομικών συμβουλών που προωθείται. Επίσης, θα προωθούσαμε μία συμφωνία σε διακρατικό επίπεδο έτσι ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να εγγραφούν σε μεγαλύτερες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελούσε μία σανίδα σωτηρίας για τις μικρομεσαίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούαν. Κυρία Σουίντορμ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το 99% της απασχόλησης στη χώρα μου είναι από τις ΜΜΕ, αλλά τώρα με την ε, ύφεση έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ε, ε παρόλες τις πρωτοβουλίες δεν ε, βοηθούνται τη σήμερον ημέρα και με το άσχημο οικονομικό κλίμα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επειδή ο χρηματοδοτικός στόχος είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στις ε, πιο αυτοχές περιοχές θα ήθελα να η Κομισιόν να ενθαρρύνει τις ε, περιφερειακές αρχές ε, να χρησιμοποιήσουν υπέρ των ΜΜΕ τα κονδύλια αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί έτσι απασχόληση και θέσεις εργασίας που θα αντέξουν στην κρίση. Ε, χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία και πιο συντονισμένη δράση. Ας το κάνουμε αυτό για να δώσουμε καινούργια κίνητρα και ερεθίσματα στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Τέλος. Ε, κυρία Γκάλ, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που θα απευθύνονται στι ΜΜΕ, θα τις καλύψουν και όλα αυτά τα θέματα τα οποία σήμερα ακούσαμε μα καταδείχνουν ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα για να μπορέσουμε τελικά να επαγρυπνούμε, να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τι ΜΜΕ, πώ θα έχουν ένα περιβάλλον ευμενέ για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ΜΜΕ. Οπότε η σημερινή κρίση μα ε, δείχνει κάποια πράγματα. Μα δείχνει ότι θα πρέπει τώρα να προσέξουμε την ε, πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Ε, πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τις ΜΜΕ να τις διευκολύνουμε διότι οι πιο καινοτόμε επιχειρήσει τώρα υποφέρουν από τι σχετικέ ε, συνέπειε, διότι θα πρέπει να δούμε το ότι θα βγούμε από την κρίση εάν βοηθήσουμε τι μικρέ επιχειρήσει. Το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα πρέπει να τι βοηθήσουμε. Πώ θα το καταφέρουμε αυτό πώς θα μπορέσουμε να τους δώσουμε ε, τα μέσα τα οποία χρειάζονται για να προχωρήσουν. Εγώ συμφωνώ με την ιδέα αυτού του τεστ για τις ΜΜΕ και ότι να, να, να συρρυκνώσουμε και να προσθέσουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Γκάλ. και ε, ευχαριστούμε και τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις και για τα θέματα που θίξατε που άκουσα με μεγάλη προσοχή και βεβαίως θα τα κοινοποιήσω όλα αυτά στο συνάδελφό μου τον κύριο Ταγιάννη. Καταρχήν, για να απαντήσω τηλεγραφικά, πολλά θέματα εφήγησαν σε σχέση με τις ΜΜΕ και μιλήσαμε για τα εθνικά οικοσυστήματα ως προς το, τη φορολογία, το, τα διοικητικά βάρη, τις ε, χρηματικές επιβαρύνσεις και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δράσουμε πανευρωπαϊκά. Θα ήθελα να πω προς την κυρία Σαρτόρη ότι όταν μιλάμε για πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι ένα κείμενο που γνωρίζετε πολύ καλά, τώρα βρίσκεται στη δεύτερη ανάγνωση στο, σε επίπεδο Συμβουλίου. Ο κύριος ε, Πασκουά μίλησε για την αρμοδιότητα των κρατών μέλων και η κυρία Σουίνμπερν μίλησε και πάλι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τις οποίες πρέπει να διευκολύνουμε. Οι κύριοι ε, Μπρόνς, ε, Ρινάλντι, ε, Ριβέρα, Προβέρα μάλλον και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν εκ νέου σε αυτό που προανέφερα, δηλαδή τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Όταν μιλάμε για τους κανόνες της Βασιλείας, Βασιλεία 3 για τις ε, κοντά στις 2.000 ευρωπαϊκές τράπεζες, εάν εφαρμόσουμε τους κανόνες όπως ορίστηκαν από τους G20, θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της εκ νέου κεφαλαιοποίησης στον κοινωνικό ιστό. Και ο κύριος Ταγιάννη θα προβεί σε μία ανακοίνωση επί του θέματος αυτού στις 9 Νοεμβρίου. Θα ήθελα να πω στον κύριο Βάτσον και στον κύριο Ρούμπιχ ότι και εγώ μίλησα για έλεγχο και φορολόγηση. Ο κύριος Σεμέτα καταρτίζει μια πράσινη βίβλο που θα παρουσιάσει κατά τα τέλη του 2011 ε, μιλώντας για αυτό το θέμα της απλούστευσης της ε, πλαισίως του ΦΠΑ, ιδιαίτερα ως προς τις διασυνοριακές υποχρεώσεις. Η κυρία Μέρκης μίλησε για μια δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες ε, που δεν προβαίνουν σε πτωχεύσεις χωρίς να συνίσταται λόγος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα υψηλό ποσοστό πτωχεύσεων είναι απατηλές πτωχεύσεις και η διαδικασία ε, αποκατάστασης είναι μία μακροχρόνια διαδικασία. Γι' αυτό χρειάζονται τουλάχιστον, μάλλον υπάρχει ένα όριο τριών ετών για τους υγιείς και έντιμους επιχειρηματίες έτσι ώστε να μπορέσουν να ξαναρχίσουν. Και η Επιτροπή θα δει τι πρόοδος έχει επιτελεστεί. Αυτό θα ήθελα να πω στην κυρία Μέρκης. Προς τον κύριο Κέλλη θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια του Single Market Act μιλώ για κινητικότητα του κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου στο Μόναχο συνεδριάσαμε και μιλήσαμε για τις μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται αυτή τη χρηματοδότηση. Η κυρία Τόγια και η κυρία Χάνσλικ έθιξαν το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών και της σωστής εφαρμογής αυτής της οδηγίας, ο κύριος Ταγιάννη έκανε έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές. Θα ήθελα να πω στον κύριο Λούχαν και θα επανέλθω, αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο. Με τον κύριο Ταγιάννη και τον κύριο Σεμέτα προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε εξειδικευμένη νομοθεσία για τις ΜΜΕ και μιλήσαμε για τις δημόσιες συμβάσεις όπου θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, προσβασιμότητα. Ε, κύριε Νίκολσον, προσπαθούμε να άρουμε την γραφειοκρατία και αλλού, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, και στις Βρυξέλλες υπάρχει γραφειοκρατία και προσπαθούμε ανανομοθετική πράξη να μειώσουμε το γραφειοκρατικό φόρτο σε εθνικό επίπεδο. Οι κύριοι Νίκολσον και Γκάλαχερ ε, μίλησαν για αυτό το τεστ ΜΜΕ, εμείς προβαίνουμε σε αυτή τη δοκιμή ΜΜΕ σε κάθε κράτος μέλος για να δούμε πόσο μπορούμε να το φέρουμε σε αίσιο πέρας. Ο κύριος Μπουτιχόφερ μίλησε για τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων δηλαδή την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών γενικών διευθύνσεων, καταβάλουμε ε, μεγάλες προσπάθειες με τους συναδέλφους Κουίν και Ταγιάννη. Θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, κύριε Μπουτικόφερ, για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την ε, καλύτερη προσβασιμότητα σε κονδύλια έρευνας. Ως προς την τυποποίηση, η πρόταση Ταγιάννη συζητείται και μπορώ να σας πω ότι μέσω αυτών των ε, συνεργασ... αυτής της συνεργασίας για την τυποποίηση προσπαθούμε να μην γίνονται διακρίσεις. Ο κύριος Κάρινς ρώτησε από πού θα προέλθει η ανάπτυξη. Όταν δούμε τη σημασία των ΜΜΕ, το 99% του οικονομικού ιστού, γνωρίζουμε ότι οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να προσαρμοστούν πολύ καλύτερα για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και θα είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα των συνόρων, αλλά χωρίς αφελείς σκέψεις. Γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό το μέσο αμοιβαιότητας ως προς τις δημόσιες συμβάσεις στις μεγάλες περιφέρειες. Πολλοί μίλησαν, μάλλον ε, ένα συνάδελφό σας μίλησε για την επανεθνικοποίηση. Εγώ ε, διαφοροποιούμε, γιατί διαφορετικά θα κατακαιρματιστεί η ενιαία αγορά. όταν πάτε στις ΙΠΑ ή στην Κίνα βλέπετε ότι μας σέβονται επειδή έχουμε μία μεγάλη ε, αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών και 22 εκατομμυρίων επιχειρήσεων. Ας μην συρρυκνωθούμε εκ νέου. Η κυρία Μπασέσκου μίλησε για κονδύλια κατάρτισης. Νομίζω ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια, δυστυχώς. Επειδή μίλησα λοιπόν για την ανάπτυξη, θα ήθελα να πω, κύριε Ταγιάννη, ότι, ε, ότι με τον κύριο Ταγιάννη εργαζόμαστε επί ενός θέματος που δεν είναι και τόσο εύκολο. Παλιά το να μιλάει κανείς για βιομηχανική πολιτική ήταν κάτι το πολύ παράτολμο. Νομίζω ότι μετά την ΕΚΑΧ θα πρέπει να, να δούμε τι βήματα κάναμε μέχρι το Airbus με βάση μεακούς με βάση συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς, δηλαδή τομεακή προσέγγιση. Μας ενδιαφέρει η βιοτεχνολογία, η δημόσια υγεία, οι μεταφορές. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα δηλαδή να είμαστε ανεξάρτητοι ως Ευρωπαίοι και να μην εξαρτώμαστε από προϊόντα ή αγαθά που παράγονται αλλού. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να είναι υποχείριο των άλλων. Χρειαζόμαστε ε, υπηρεσίες. Πρέπει να παραμείνουμε παραγωγή, να μην αγοράζουμε προϊόντα που παρασκευάζονται ή κατασκευάζονται αλλού. Γι' αυτό, και το λέω προσωπικά, ε, πιστεύω ότι με τον κύριο Ταγιάννη θα αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες για τη βιομηχανική πολιτική. Ο κύριος Σβάμπ γνωρίζει πολύ καλά την εργασία μας αυτή και η έκθεση Γκρές ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Επειδή σας ενδιαφέρει η τύχη των μικρών επιχειρήσεων, θα ήθελα να δείτε αυτούς τους ε, πίνακες του Single Market Act. Τον δείχνει τον πίνακα ο Επίτροπος. Είδαμε 12 μοχλούς, εντοπίσαμε 12 μοχλούς και 50 προτάσεις, εκ των οποίων η καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα ε, Τεχνίας κατέχουν σημαντική θέση και θα προσπαθήσουμε στην αρχή του επομένου έτους να μπορέσουμε να προβούμε σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι καθοριστικής σημασίας έτσι ώστε να έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ευκαιριών και όχι συρρήκνωσης. Ξέρετε ότι δεν είμαι υπέρ θεωρητικών πλαισίων. Ως προς τις ΜΜΕ θεωρώ ότι θα πρέπει να τους διευκολύνουμε τη ζωή, να υπάρχει καινοτομία, κινητικότητα, σωστή φορολόγηση και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμφιλιώσουμε τις ΜΜΕ με τη μεγάλη αγορά, διότι ε, θα θέλαμε αυτή η αγορά να μην αφορά μόνο τους μεγάλους. Και ελπίζω να το ε, συμμεριστείτε και εσείς αυτό. Αυτό ήθελα να πω και στην κυρία Ντελκαστήγιο Βέρα και στον κύριο Σουβάπ. Υπάρχει ένας ε, διαδικτυακός τόπος για τις ΜΜΕ και για την κατάρτισή τους και θα επανέλθουμε με τον κύριο Ταγιάννη επί του θέματος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία σαν να επρόκειτο για μία σύμβαση ΜΜΕ Ευρώπη. Αυτά να ήταν τα δύο συμβαλόμενα μέρη δηλαδή. Είμαι πεπισμένος ότι έτσι θα βοηθήσουμε αρκούντος τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε Μπαρνιέ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση σε αυτό το σημείο. Το επόμενο σημείο είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού σύμφωνα με το